πρέπει να έχει μια αυτάρκεια στον τομέα αυτό. Και δεν μπορεί κανείς λοιπόν να ξεχάσει αυτή τη βασική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> Σας ευχαριστώ. Κυρία Κιώστιγκερ, μπαίνουμε στην οφθαλμοθερευτική διαδικασία. Η κυρία Ρόιτοβα έχει το λόγο πρώτα.